Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξαναβλεπόμαστε και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα πάλι. Καλώς ήρθατε κι εσείς και ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, που θα μας κάνουν τη διερμηνία σε αυτή τη συνεδρίαση Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Φόρουμ θα βρείτε στο τραπέζι μπροστά ε, ζάχαρη από τη Ρεϊνιό, που είναι η γενέτηρά μου. Και για την περισμένη φορά είχαμε πολύ έντονε εργασίε και είχαμε εξαντληθεί. Γι' αυτό σκέφτηκα να βρω κάποιο καύσιμο να μα δώσει ενέργεια για να κρατήσουμε ακμαία τη δύναμή μα καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών μα. Γι' αυτό και σα μοιράσαμε ζάχαρη από τη Ρινιό. Ζάχαρη, άλλωστε, η παραγωγή ζάχαρη είναι από τους βασικούς κλάδους στα νησιά αυτά. Και στην αντιπροσωπεία μας θα μιλήσουμε για αυτά τα νησιά. Γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και θα ασχοληθούμε κυρίως με το θέμα της καταπολέμησης ή του μετριασμού των κλιματικών αλλαγών που επηρεάζει άμεσα τα νησιά παντού στο πλανήτη. Και θα ήθελα να μιλήσουμε εδώ ελεύθερα για το σενάριο που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας αυτή τη στιγμή και που δεν αγγίζει μόνο τα νησιά του Καριφόρου. Αυτό είναι ένα από τα δύο σημεία τη ημερήσια διάταξη. Το δεύτερο σημείο είναι η πορεία των διαπραγματεύσεων για την συμφωνία μετά το Κοτονού. Και θα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μα η συντονίστρια των χωρών του Καριφόρουμ, η εξοχότατη Σέιλα Σίλι Μόντε, που είναι πρέσβυρα της ε, Τζαμάικα. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και τον ε, πρέσβη του Μπελίζ. Και σε αυτή τη βίντεο διάσκεψη που είχαμε την περασμένη φορά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε αρκετά και σήμερα πιστεύω θα έχουμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση. Η διαδικασία μας υποχρεώνει να εγκρίνουμε πρώτα τα πρακτικά της συνεδρίασης της 18 Δεκεμβρίου του 2019. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή αισθάσεις από πλευρά σας, θα θεωρηθούν συγκεκριμένα τα πρακτικά. Και περνάμε στο κυρίως θέμα της σημερινής μας συζήτηση, τις κλιματικές αλλαγές. Ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, αλλά που πλήττει κυρίως ιδιαίτερα και γίνεται πολύ πιο αισθητό στα μικρά νησιωτικά κράτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, έχει υιοθετήσει μια πολύ φιλόδοξη νέα πράσινη συμφωνία, το New Green Deal που λέμε, και που έχει στόχο να μεταμορφώσει τις οικονομίες μας με απότερο σκοπό να γίνουμε ουδέτεροι από άποψη σου άνθρακα μέχρι το 2050. Γι' αυτό όμω θα πρέπει να αναθεωρούμε συνεχώ και να επανεξετάζουμε τον τρόπο παραγωγή μα, τον τρόπο κατανάλωσής μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχουμε εμπορικές συναλλαγές με τους εταίρους μας και με τους εταίρους ε, του Κάρι Φόρουμ. Έχουμε πολλούς ε, καλεσμένου σήμερα που θα μας κάνουν μια σύντομη επισκόπηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή της Καραϊβικής. Και έχω την ιδιαίτερη χαρά να καλωσορίσω τον δόκτωρα Δίλαν Βερνό, που είναι πρέσβης, όπως σας είπα, του Μπελίζε. Εξοχότατε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Άλλωστε, η χώρα σας ασκεί την Προεδρία της ΑΟΣΙΣ, της Συμμαχίας Μικρών Ισιωτικών Κρατών, που συγκεντρώνει 44 χώρες, είτε μικρές ισιωτικές χώρες, είτε παράκτιες ε, χώρες χαμηλού υψομέτρου. Και η συμμαχία αυτή έχει πρωτοστατήσει στις εργασίες του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Επίσης δίπλα σας έχουμε την κυρία Λένη Ισμαέλ, πρώην πρέσβυρα των χωρών της Ανατολικής Καραϊβικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρμόδια για τις πολιτικές ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό ε, Κέντρο Ερευνών για τη διαχείριση των αναπτυξιακών πολιτικών. Θα δώσω λοιπόν σε όλους τους καλεσμένους μας το λόγο για να μας φωτίσουν με την εμπειρογνωσία τους. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Δίλαν Βένον, τον πρέσβη του Μπελίζε και να τον ευχαριστήσω και να τον καλωσορίσω και πάλι θερμότατα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εσάς και την αντιπροσωπεία σας για την πρόσκληση που μας κάνατε να έρθουμε εδώ και να σας μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι υπαρξιακή προτεραιότητα για τις χώρες Καριφόρουμ. Όπως είπατε, με καλέσατε για να κάνω μιας, κάποιες παρατηρήσεις, να σας παρουσιάσω τις απόψεις μας γιατί ασκούμε την Προεδρία της ΑΟΣης αυτή τη στιγμή, της συμμαχία των Μικρών Ισιωτικών Κρατών, στο οποίο συμμετέχουν 16 κράτη-μέλη και του Καριφόρου. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Μπελή είναι ε, η πρώτη παράκτια χώρα χαμηλού υψομέτρου που ασκεί την Προεδρία του Συμμαχία ΑΟΣης. Όπως ξέρετε, οι χώρε μα. Ε, ήταν πρωτοπόρε στις κλιματικέ δράσει, γιατί βιώνουμε στο πετσί μα ε, και είμαστε στην πρώτη γραμμή ε, των χωρών που επηρεάζονται από αυτέ τι κλιματικέ αλλαγέ. Και παρόλο που η ομάδα μα συμβάλλει με λιγότερο από 1% στι παγκόσμιε εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, κάνουμε ό,τι μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές μας αερίων του θερμοκηπίου και να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να έχουμε πιο πράσινη και κοινωνία και οικονομία. Και μάλιστα πρωτοστατούμε στην αναθεώρηση των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών μας, προκειμένου να δώσουμε έμπνευση και σε άλλες χώρες ε, να αναβαθμίσουν και αυτές τις εθνικές, εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους. Πάντως, ε, οι χώρες καριφόρμ, όπως ξέρετε, είναι αυτές που υφίστανται το μεγαλύτερο κίνδυνο από τις κλιματικές αλλαγές. Βέβαια, είχαμε ήδη πολλές απώλειες και ζημιές σε όλα τα κράτη του Καριφόρουμ και έχουμε παρόλα αυτά τεράστιες προκλήσεις ε, για να προσαρμοστούμε στη νέα κατάσταση και να αποτρέψουμε τις ε, περιβαλλοντικές καταστροφές. Ήδη βιώνουμε μια κλιματική ανασφάλεια που έχει τεράστιες επιπτώσεις σχεδόν σε κάθε πτυχή της κοινωνίας, ε, της οικονομίας μας, αλλά ακόμη και της μετανάστευσης. Και εν ώψη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη Καριφόρουμ, και δεδομένη εγγενή τροτότητα και ευπάθειά μα που επιδεινώνεται από τι επιπτώσει των κλιματικών αλλαγών, έχουμε προκλήσει που περιλαμβάνουν περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, περιορισμένη παραγωγή λόγω του μικρού μα μεγέθου, τεράστιο χρηματοπιστωτικό άχθό λόγω του χρέου μα και επιστηστική ανασφάλεια. Μάλιστα είχαμε τον ε, τυφώνα Ντόριαν του 2019 που χτύπησε τις Μπαχάμες και μας υπενθυμίζει τις πολλαπλές ευπάθειες που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας. Μόνο και ένας τυφώνας Ντόριαν μπορεί στην περιοχή να εξαφανίσει ε, το ΑΕΠ μιας χώρας. Είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα παντού στην περιοχή. Είχαμε και ανοβρίες, πλημμύρες, διάβρωση των ακτών. Και μάλιστα οι χώρες της Καραϊβικής αναγνωρίζουν και εκτιμούν ιδιαίτερως τις δεσμεύσεις και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα αφήσω το λόγο ε, στους συναδέλφους από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα για να μας παρουσιάσουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε μια πιο δυναμική και αναβαθμισμένη κλιματική φιλοδοξία. Θα θυμάστε την ε, ειδική έκθεση της ομάδας της Επιτροπής του ΟΗΕ για το κλίμα, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη κατά δύο βαθμούς θα οδηγήσει σε τεράστιες ζημιές και απώλειες σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Επίσης, θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ στις δράσεις που έχουμε κατά προτεραιότητα ανάγκη. Βέβαια, εμείς θέλουμε φιλόδοξες δράσεις για μετριασμό και προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και να προσαρμοστούμε και να δημιουργήσουμε μια θεκτικότητα απέναντι στις θεομηνίες και τις φυσικές καταστροφές. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια αναθεωρημένη συμφωνία σχέση για να έχουμε ε, ε, λιγότερες εκπομπές, λιγότερες ζημίες, να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενισχυμένη διεθνή συνεργασία και χρηματοδότηση στοχευμένη σε συγκεκριμένα θέματα. Και γι' αυτό ε, είναι σημαντικό να συνεχιστούν ε, οι υποσχέσει χρηματοδότηση του Ταμείου για την Προσαρμογή στι Κλιματικέ Αλλαγέ. Επίση, θέλουμε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση σε επιδοτήσει και σε ε, δανεισμό με ευνοϊκού όρου. Και μάλιστα, ε, εμεί ε, έχουμε αναβαθμιστεί και έτσι έχουμε χάσει την επιλεξιμότητά μα από την επίσημη βοήθεια. Και μερικέ χώρε αντιμετωπίζουμε ανάγκες επιβίωση, Μάλιστα πολλές φορές επειδή έχουμε προφίλ ψηλού κινδυνού έχουμε εκτοπιστεί και από τις χρηματοπιστωτικές ε, αγορές. Παρ' όλα αυτά είμαστε πρωτοπόροι στην ε, πρόθεση μιας διεθνούς σύμβασης ε, για την διαφύλαξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Έχουμε κοινούς στόχους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χώρες ΑΚΕ για την περίοδο μετά το Κοτονού είναι μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουμε την εταιρική μα σχέση για ενισχυμένες κλιματικές δράσεις. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής ε, επηρεάζει κυρίω τα μικρά νησιωτικά κράτη και γι' αυτό ε, προτείνουμε το σχετικό πρωτόκολλο να επισυναυθεί και σίγουρα Θέλουμε το νέο πρωτόκολλο και νέα συμφωνία να ευοδοθούν, να τελεσφορήσουν και αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά από τα μέσα που θα διατεθούν για την αναπτυξιακή συνεργασία. Και εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διδραματίσει κέριο ρόλο. Θα ήθελα λοιπόν να συνεργαστούμε κύριε Πρόεδρε και με εσά και με τους συναδέλφου σα. και θα πρέπει το θέμα των κλιματικών αλλαγών και την ευπάθεια αυτών των χωρών να το θέσουμε ως κοινό στοιχείο του προγραμματός μας. Και παρόλο που είμαστε δύο διαφορετικές περιοχές του κόσμου, είμαστε ένας λαός, μία ανθρωπότητα, ένας πλανήτης με κοινό πεπρωμένο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, εξοχότατε που μας ε, περιγράψατε και τις, ε, μας δώσατε τη μαρτυρία σας για την πραγματικότητα και μας μεταφέρατε τις εμπειρίες σας για το τι ζουν οι χώρες ε, του Κάριφόρν και πολύ σωστά τονίσατε τον πολύ ευάλωτο χαρακτήρα αυτών των περιοχών απέναντι στον οποίο φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αρκεστεί ε, στις απαιτήσει που προβάλλουμε σήμερα και τις οποίες πρέπει να πετύχουμε με την Πράσινη Συμφωνία αλλά είναι απαραίτητο να εξευρεθούν λύσεις αν αντιμετωπιστεί η απορρίθμιση του κλίματος. Προτείνω λοιπόν να συνεχίσουμε την ανταλλαγή εμπειριών και αυτή τη φορά θα δώσω το λόγο στην δόκτωρα Λέν Ισμαήλ. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που είστε εδώ. Όποιοι ήρθαν τώρα να πω ότι είστε τέος πρέσβυρα των κρατών της Ανατολικής Καραϊβικής ε, και είστε ερευνήτρια σε θέματα πολιτικής, αναπτυξής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσω μαζί σας σήμερα ένα από τα πιο ακαθόδη ζητήματα των καιρών μας, που είναι η εκτακτή κλιματική κατάσταση. Έχω λίγο χρόνο, θα ήθελα λοιπόν να περιστώ σε λίγες σκέψεις. Πρώτον, η κλιματική αλλαγή είναι ένα μόνο παράγων που συνεισφέρει στον ευάλωτο χαρακτήρα των μικρών νησιωτικών αναπτυξιακών κρατών. Απλά έχει τεράστιο μέγεθο, είναι συστημικού χαρακτήρα λόγω του μεγέθου των νησιών και υπαρξιακή φύσεω. Δεύτερον, τα μικρά νησιωτικά κράτη τη Καραϊβική έχουν πετύχει Ψηλά επίπεδα ανθρώπινη ανάπτυξη, με ξέρει την ΑΕΤ, είναι χώρε μέσω εισοδήματο. Είναι πολύ σίγουρα αξιοζήλευτο αυτό το που έχουν πετύχει, αλλά κρύβει και πολλέ αλήθειε ότι έχουμε συνεχή φτώχεια, σταθερή φτώχεια, 30% τουλάχιστον του πληθυσμού, ε, όταν ιδίω ε, στο νοικοκυριό είναι η γυναίκα είναι πολύ ευάλωτα. Έχουμε πολύ χρεωμένε χώρε, πολύ μεγάλη ανεργία που φτάνει και το 40%. Επίση, υπάρχουν και εγγενεί ασθενείς ε, ε, τροτότες, οι οικονομίες μας είναι μικρές, ανοιχτές και πάρα πολύ εκτεθειμένες στις παγκόσμιους κραδασμούς της αγοράς. Χτυπήθηκαν πολύ βαριά από την επιστηστική κρίση και την κρίση του πετρελαίου το 2007 και την κατάρρευση των χρηματοπιστών αγορών το 2008. Και η κατάσταση αυτό, το μέσο εισόδημα που έχουν αυτές οι χώρες δεν τους έχει δώσει οικονομική ανθεκτικότητα. Ε, υπάρχει οικονομική και κοινωνική ε, αδυναμία ε, ρευστότητα και ε, εύθραστη είναι η κατάσταση μέχρι το επόμενο αυτό σοκ. Επίσης είχαμε πολλές φυσικές καταστροφές, 10 τυφώνες, 3.600 θανάτου, 290 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια ζημιών που κατέστρεψαν πάρα πολλά από όσα είχαμε πετύχει στη Βόρεια Καραϊβική και το 2017 έτσι έγινε η χειρότερη εποχή των παράκτηων τυφών στην ιστορία της Καραϊβικής. Έχουμε μικρό ποσοστό δημόσιων υποδομών που όμως τώρα ε, καλύπτεται από τις ε, ε, ασφαλίσεις που δεν καλύπτουν όμως τους απλούς πολίτες, τους κατοίκους που πολλές φορές έχουν χάσει τα σπίτια τους, που έχουν χάσει τα πάντα. Η επίτευξη λοιπόν των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για τα μικρά νησιωτικά κράτη και η ανοικοδόμηση δεν είναι μόνο μια απλή πρόκληση. Πού να στραφούμε. Πρέπει να βρούμε λύσεις στα πιο επιζήμια αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής που και αυτό υπερβαίνει σίγουρα τις δυνατότητες ενός μονοκράτους. Ε, ε, δεν μπορεί να το διχειριστεί κάποιο κράτος μόνος του. Έχουμε συμφωνίες που βασίζονται στις αρχές του πολυμερού συστήματος αυτή είναι η μόνη ελπίδα, παρά το ότι έχουν διαβρωθεί κάπως προσφάτως. Χαιρετίζουμε την διάταξη, ε, μάλλον την παγκόσμια ηγετική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το πράσινο σύμφωνο, ε, που είναι κάτι θετικό για να βάλουν οι Ευρωπαίοι τα, του οίκου τους σε τάξη, αλλά έχουμε και πολλές άλλες σημαντικές προκλήσεις και επίσης θα είναι πολύ δαπανηρή μετάβαση σε ουδέτερος προς τον άνθρακα συστήματα. Υπάρχουν επίσης πολλές πρωτοβουλίες όπω είναι παραδείγματο χάρη η Παγκόσμια Συμμαχία για την Κλιματική Αλλαγή. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ε, η προσαρμογή θα απαιτήσει, έχει κάποια τεχνικά και οικονομικά όρια ε, και θα απαιτήσει πολύ σκληρέ επιλογέ. Ε, Επίση, πρέπει οι χώρε, οι μικρέ νησιωτικέ χώρε Καραϊβική, να αναπτύξουν οικονομικά αποθέματα ώστε να μπορούν να είναι ανθεκτικέ, να έχουν ένα μαξιλάρι, αν θέλετε, για να αντιμετωπίσουν καταστροφικά ε, γεγονότα. Δύσκολο όμω να υπάρξουν πλεονάσματα από τι τρέχουσε συνθήκε. Πώ μπορούμε να το διαχειριστούμε. Εύκολε λύσει δεν υπάρχουν. Χρειάζονται πολιτικέ και εταιρικέ σχέσει ανανεωμένε. Ε, μάλλον τρει τελευταίε γρήγορε θέσει. Πρέπει να δούμε με διαφορετικό πρίσμα την ανάπτυξη. Δεν είναι ένα γραμμικό οικοδόμημα όπου οι χώρες πηγαίνουν από ένα πιο χαμηλό σε ένα πιο υψηλό επίπεδο ανάπτυξη. Είναι μια κυκλική διαδικασία. Οι χώρες κάνουν βήματα προς τα εμπρός αλλά και βήματα προς τα πίσω. Αρκεί μια καταστροφή, φυσική καταστροφή για να χαθούν κέρδη ε, δεκαετιών. Η οικοδόμηση οικονομικής ε, αντοχής ε, για τις χώρες αυτές απαιτεί οικονομική ανάπτυξη και ένα παραδιαθέσιμο εργαλείο είναι η οικονομική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Κάρι Φόρουμα. Εννέα χρόνια μετά βέβαια βλέπουμε ότι δεν έχουν αποκρισταλωθεί τα ωφέλη και τα κέρδη για τις περισσότερες χώρες Καραϊβικής. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η εταιρική σχέση να επανεξεταστεί. Το περιφερειακό πρωτόκολλο ε, Επίση ε, που διαπραγματεύεται τη μετά το κοτονού κατάσταση είναι και αυτό μια άλλη ευκαιρία. Επίση, το λεγόμενο blending είναι ένα πολύ χρήσιμο οικονομικό εργαλείο αλλά θα πρέπει στι μικρέ ε, κοινωνίε οι πολιτικέ να είναι προσαρμοσμένε για να φτάσουν ακριβώ στου πλέον ενδεεί. Θα πρέπει να του βοηθήσουν να επισκευάσουν φτωχικέ κατοικίε, πρέπει να στηρίξουν προγράμματα μετεγκατάσταση, απαιτούνται προσιτά οικονομικά ασφαλιστικά συστήματα θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για να κλεισεί το χάσμα μεταξύ των πολιτικών Αφενό και των αποτέλεσματο που έχουν επιτόπου. Τέλο, έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ομάδα των 8 και την ομάδα των 20, την εταιρική σχέση με τι χώρε ΑΚΕ, ε, τις ΑΚΕ μαζί με την ομάδα των 77 και την Κίνα. Όλοι μα διμερό ή πολυμερό, θα πρέπει να αναλάβουμε και να ασκήσουμε την πολιτική ευθύνη που συνοδεύει την κλιματική διπλωματία. Πρέπει να καταρτιστεί ένα θεματολόγιο για την αλλαγή. Θέλουμε τους στόχους ε, και τις οικονομικές δεσμεύσεις ε, της Συμφωνίας των Παρισίων να τις μεταφράσουμε σε συγκεκριμένες ενέργειες, σε συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές τουλάχιστον έχουμε το μονοπάτι στην Γλασκόβη και την COP26. Ε, ελπίζουμε αυτό να μην στρωθεί με ε, ακόμα πιο πολλές κενές υποσχέσεις που θα παραβιαστούν και από ε, πάρα πολλές φιλοδοξίες που δυστυχώς κάποιος θα τις παραμερίσει πάλι και να περιμένουν επόμενη διάσκεψη συμβαλωμένων. Πολλά χρειάζεται ο πλανήτης, δεν πρέπει να περιμένει πια πέρασε ώρα για τα λόγια. Ε, πρόεδρο, συμφωνώ απόλυτα. Ο πλανήτη δεν έχει χρόνο να περιμένει ε, και να γνωρίζετε ότι στην αντιπροσωπεία μα έχουμε μέλη και τη Επιτροπή Ανάπτυξη που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα ζητήματα ε, τη οικονομική ε, ευάλωτη κατάσταση των χωρών που μα εξηγήσατε εδώ. Έχουμε επίση μέλη και τη Επιτροπή ΣΥΝΤΑ Διεθνού Εμπορίου. Επομένω, η έκκλησή σα για τη ε, διαπραγμάτευση και τη συζήτηση για τι συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου θα εισακουστούν. Θα συνεχίσω το γύρο ανταλλαγής εμπειριών με τον κύριο Μανιουέλ Καρμόνα Γέρμπα από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Κλίμα. Τρία λεπτά έχετε παρακαλώ στη διάθεσή σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία. Το ένα αφορά τις κλιματικές προσωμιώσει για την περιοχή. Το δεύτερο είναι η κλιματική συνεργασία με, τη, με τα κράτη της περιοχής και το τρίτο θέμα αφορά το μέλλον και κυρίως τη νέα πράσινη συμφωνία. Καταρχήν αναφέρθηκε και από τους καλεσμένους ε, ότι υπάρχουν πολλές επιπτώσει και πέραν των τυφώνων που έχουν ρημάξει την περιοχή και αναμένεται να αυξηθούν και στην έντασή τους όπως ε, δήλωσε επανειλημμένος εκθέστης η Επιτροπή για το Κλίμα του ΙΕ έχουμε και άλλου είδους περιστατικά, όπως ε, βροχοπτώσεις και κυρίως μία ανησυχητική τάση που είναι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα pattern των βροχοπτώσεων. Επίσης, ε, αναφέρονται καλοκαίρια στην Καρεβική που θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 40-50% οι βροχοπτώσεις μέχρι τα τέλη του αιώνα. Ε, κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε αύξηση της ξηρασίας, ε, αυτή η ανοβρία θα ξηράνει το έδαφος, θα επηρεάσει τη γεωργία και εδώ μιλούμε για, μια, για ένα φάσμα επιπτώσεων, όχι μόνο για τις καταστροφικές επιπτώσεις των τυφώνων, αλλά έχουμε και άλλες επιπτώσεις από άλλα φαινόμενα. Τώρα, σε ό,τι φορά την υποστήριξη που θα δώσουμε για τη, με, τη, των κλιματικών αλλαγών στην περιοχή. Με δύο λόγια, αυτό που είχαμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου, όπως ξέρετε, είναι 5,1 εκατομμύρια για τις κλιματικές δράσεις και κυρίως για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση των, των κινδύνου καταστροφής. Σε ό,τι αφορά τη διμερή συνεργασία, πέραν το 61,5 εκατομμύριο, συγγνώμη, 61,5 εκατομμύριων, ψηφίσαμε και 300 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση και πάνω από τα μισά κονδύλια αφορούν κλιματικές δράσεις. Επίσης, το πακέτο για την αντιμετώπιση των δύο τυφώνων Ήρμα και Μαρία του 2017. Και εκεί είχαμε προσφέρει 300 εκατομμύρια ευρώ και μέτρα για την καλύτερη ανακατασκευή των κτηρίων προκειμένου να γίνει καλύτερη προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και τις προσωμιώσεις που έχουν γίνει για τις μελλοντικές καταστάσεις. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει και ο μηχανισμός, ε, επενδυτικός μηχανισμός για την Καραϊβική, με συνδυασμένη χρηματοδότηση και ήδη ένα δισεκατομμύριο έχουμε μοχλεύσει για τη βελτίωση των υποδομών για το κλίμα και για τη βελτίωση των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τι προσπαθεί να επιτύχει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλες αυτές τις επενδύσεις. Κυρίως θέλουμε να αναπτύξουμε την αθεκτικότητα της περιοχής στι κλιματικέ αλλαγέ. Κάτι που λείπει. Ε, αναφέρθηκε πόσο ευάλωτε είναι αυτέ οι χώρε ε, και πριν ακόμη από το κλιματικό ζήτημα και την εμφάνισή του. Και σίγουρα τα τροτά σημεία και ευπάθειες αυτής της περιοχής ε, επιδεινώθηκαν με τις κλιματικές αλλαγές. Έχουμε και την ε, διευκόλυνση του Καριφόρουμ από πέρυσι για να ε, στηριχθούν προγράμματα για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των ζημιών. Επίσης θέλουμε και η δημόσια υγεία και τα συστήματα δημόσιας υγείας να γίνουν αθεκτικά, γιατί είναι διαφορετικές οι προκλήσεις με την αύξηση της θερμοκρασίας και ίσως θα έχουμε κάποιες νέες προκλήσεις ε, που θα εμφανιστούν. Αυτά ήταν εν συντομία τα βασικά σημεία της αναπτυξιακής μας συνεργασίας και να πω και δύο λόγια τώρα για το μέλλον. Τι μας επιφυλάσσει η Νέα Πράσινη Συμφωνία που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι το Δεκέμβριο. Η Νέα Πράσινη Συμφωνία προσφέρει κάποιες ε, προτάσεις ε, ε, για την οικονομία. Θα πρέπει η οικονομία να αλλάξει άρθεν. Και γι' αυτό η Νέα Πράσινη Συμφωνία προσπαθεί να συνδυάσει διάφορα μέτρα και διάφορες πολιτικές και να λάβει υπόψη τις αλληλέδατες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε και κλιματικούς στόχους αμυγής, και μάλιστα πρόκειται να του αναθεωρήσουμε. Έχουμε το θέμα τη βιοπικιλότητα, την καθαρή ενέργεια, καθαρή κινητικότητα, κτίρια και υποδομές, δίκαιη μετάβαση για τι περιοχέ που θα πληγούν περισσότερο από την ανάγκη εμ, μετατροπής της οικονομίας σε πιο καθαρέ φιλοπεριβαλλοντικές μορφέ ενέργεια. Επίση, θα έχουμε δημόσιε διαβουλεύσει 4 Μαρτίου, την Τετάρτη δηλαδή, για το νέο σύμφωνο για το κλίμα με την ανάμειξη των τοπικών αρχών, τη τοπικής αυτοδιοίκησης και τη κοινωνία των πολιτών. Αυτή είναι μια σφαιρική στρατηγική ευρέω φάσματο. κάτι που χρειάζεται, γιατί αν οι κλιματικέ δράσει περιοριστούν στις αρμοδιότητε του Β Υπουργείου ή της Β κυβέρνηση δεν θα αρκέσουν. Χρειαζόμαστε διατομεακέ πολυεπίπεδες δράσεις και ε, αυτό είναι ακριβώ και το επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γέρμπα και χαίρομαι γιατί το υπενθύμησαν και οι καλεσμένοι μας αυτή η ανάγκη για μια σφαιρική προσέγγιση. Γιατί αυτή η έκτακτη ανάγκη για το κλίμα θα πρέπει να διέπει όλες μας τις παρεμβάσεις στον οικονομικό τομέα, στον κοινωνικό τομέα, στην παιδεία, παντού και πάντα. Θα πρέπει η προτεραιότητα του κλίματος να διατρανώνεται μονίμως και παντού, σε όλες τις πολιτικές μας και σε όλους τους τομείς. Αυτά και μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση τώρα. Αν θέλετε να συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψε, μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις προς τους καλεσμένους μας. Ο Μάρκ Ταραμπέλα πρώτος. Ακούσαμε για τον αρνητικό ενδείκτυπο που θα έχουν οι κλιματικέ αλλαγέ στα νησιά και σκεφτόμαστε κυρίω τον Ειρηνικό, τα νησιά του Ειρηνικού. Εξού και το ενδιαφέρον αυτή τη συνεδρίαση. Γιατί από ό,τι ακούσαμε, αντίκτυπο θα υπάρξει και για τα νησιά τη Καραϊβική και όχι μόνο για τα νησιά του Ειρηνικού. Δεδομένη τη σοβαρότητα, τη ένταση και τη μεγαλύτερη συχνότητα των άστατων καιρικών φαινομένων και των ακραίων φαινομένων όπω οι τυφώνες Πέραν τούτου, σε κάποια νησιά, ίσως σε μερικά περισσότερα από ό,τι σε άλλα, σας επηρεάζει και η πιθανή άνοδος της στάθμης των υδάτων στους ωκεανούς. Οι κάτω είναι η χώρα που κατεξοχήν είναι καλύτερα προετοιμασμένη με την άνοδο και των φραγμάτων για να αντιμετωπίσουν αυτή την άνοδο της στάθμης των υδάτων. Εσείς επηρεάζετε από αυτή την άνοδο της στάθμης των υδάτων, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω καλά την κατάσταση σε όλα αυτά τα νησιά. Ευχαριστώ τον Μάρκ Ταραμπέλα. Σίγουρα το Καριφόρουμ θα είναι μια καλή ευκαιρία να εξοικειωθούμε καλύτερα με όλα αυτά τα νησιά και του Ατλαντικού ωκεανού και της Καραϊβικής ιδιαίτερος. Δεν ξέρω αν οι διαπρεπείς καλεσμένοι μας ε, θα ήθελαν να απαντήσουν ε, για την απειλή που συνιστούν ε, συνιστά η άνοδος της στάθμης του ύδατος για τα νησιωτικά κράτη και τα παράκτητα κράτη της Καραϊβικής και του Καριφόρου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι όλα τα νησιά θα πληγούν από την αύξηση τη των υδάτων ε, στην Καραϊβική. Ορισμένα νησιά είναι και ηφαιστειακά, ηφαιστειογενή, που σημαίνει ότι υπάρχουν τμήματα των νησιών που δεν θα πληγούν, όμως οι παράκτιες ε, περιοχές εκτογραμμένων των νησιών θα επηρεαστεί. Θα υπάρξουν επίση αλλαγές ε, και στα παράκτια οικοσυστήματα και στις κοραλιογενείς περιοχές, ε, τις ε, αμοθήνες και όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ και τους φυσικούς πόρους από τους οποίους εξαρτώνται οι κάτοικοι των νησιωτικών αυτοκρατών και οι υποδομές σχεδόν στο σύνολό τους σε όλα τα νησιά είναι παράκτιες και το δικό δίκτυο, οι αερολιμένες, τα νοσοκομεία, οι κοινωνικές δομές είναι κοντά στις ακτές, όλα όλα αυτά κινδυνεύουν. Ε, ο Ειρηνικός, ε, πολλά νησιά του Ειρηνικού ήδη ε, βυθίζονται. Έχουμε χάσει αρκετά κομμάτια θα έλεγα του, του, των πόρων και μεγάλο μέρος των πόρων στα νησιά χαμηλού ψωμέτου. Είναι πάντως μια καταστροφή που διαγράφεται σχεδόν για το σύνολο των νησιών της περιοχής. Ευχαριστώ. Αυτό εξοχώτης. Ναι, πολύ σύντομα να προσθέσω πως από τα 16 κράτη-μέλη του Καριφόρουμ, τα τρία δεν είναι νησιά, έχουν όμως νησιά ε, και χαμηλαίου ε, μέτρου παράκτιες ε, περιοχές που επηρεάζονται σίγουρα. Για τις υποδομές θα ήθελα να πω κάτι. Ένα μέρος Ε, της μελλοντικής εταιρικής σχέσης ε, μας θα είναι και η μεταφορά τεχνολογίας ε, εκεί που θα μπορούσε η αντοχή, η αθεκτικότητα να δημιουργηθεί με δατοφράκτες για παράδειγμα ή με, με άλλα τέτοια μέτρα και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ. Ξεχότατε να υπενθυμίσω τον Μπελίζε αυτή τη στιγμή προεδρεύει τη Συμμαχία των Μικρών Νησιωτικών Κρατών και επειδή μιλούμε για περιβάλλον γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο νησιωτικό πλαίσιο πέραν ε, της καταπολέμησης της του κλίματος υπάρχει και αυτό το γενικότερο πλαίσιο των θεμάτων που άπτονται του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή, εν τέλει, ε, σε ένα μικρό εδαφο ε, σε ένα νησί, πώς μπορούν να αναπτυχθούν οι καθημερινές πρακτικές ε, για να οδηγήσουν σε περισσότερο σεβασμό του περιβάλλοντος μέσω της κυκλικής οικονομίας. Ε, στη συμμαχία σας υπάρχουν ε, τέτοιου είδους συζητήσεις, αναζητούνται, έχουν εξευρεθεί λύσεις. Υπάρχει και εδώ η ανάγκη να απευθύνουμε έκκληση για συνεργασία και συγκεκριμένα εσείς να απευθύνετε έκκληση για συνεργασία με εμάς στην Ευρώπη. Ακούστε, Θέλω να πω ξεκάθαρα εδώ ότι ο πρόεδρος ε, είναι και πρέσβης της Νέας Υόρκης που ε, θα μπορούσε να απαντήσει. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι σε ό,τι αφορά τα μικρά νησιωτικά κράτη και δι της Καραϊβικής, σίγουρα υπάρχουν οικονομικά ζητήματα και υπάρχει σαφής διασύνδεση μεταξύ του αντίκτυπο που έχει στις οικονομίες μας η κλιματική αλλαγή και της ανάγκης να βελτιώσουμε την οικονομική μας ανθεκτικότητα. Ε, ορισμένα μέτρα τα λαμβάνουμε ήδη από μόνοι μας, λόγω του μικρού μεγέθους και των περιορισμένων επιλογών ε, σε ό,τι αφορά την οικονομική παραγωγικότητα, έχουμε τεράστιες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Όμως, το παλεύουμε και το παλεύουμε και με την υποστήριξη και ήδη έχουμε την εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το θέμα είναι πώς μπορούμε να την βελτιώσουμε την εταιρική αυτή σχέση, ιδίω για να έχουμε περισσότερη οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο για τις ε, ομιλίες σας, αλλά και για τις απαντήσεις που δώσατε. Και πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο, που φυσικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το πρώτο, γιατί αναφερθήκατε για τη συμφωνία μετά το Κοτονού. Θα επανέλθουμε δηλαδή στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να πω ότι αυτά που είπατε έχουν θεμελιώδη σημασία. Καταρχήν, κάθε φράση που προφέρατε έχει τη βαρύτητα και τις γνώσεις της εμπειρογνωσίας σας, αλλά και της ε, κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε και δείχνει το είδος ε, του αγώνα που έχουμε να δώσουμε για να μετριάσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Και πραγματικά είναι τεράστια η αλληλεπίδραση μεταξύ ημών και ημών, μεταξύ όλων των κατοίκων του πλανήτη. Θα πρέπει λοιπόν από κοινού να αναζητήσουμε τις λύσεις και μαζί θα πρέπει να αναλάβουμε και να αναβαθμίσουμε τις πρωτοβουλίες μας, να αναβαθμίσουμε την καινοτομία, γιατί χρειαζόμαστε την καινοτομία και τον εταιρισμό και να προωθήσουμε τα ταλέντα που έχουμε παντού ώστε να συνεργαστούμε, γιατί αυτό είναι το πνεύμα που θα θέλαμε να διέπει τη Συμφωνία του Καριφόρουμ. Δηλαδή, οι λύσεις που υπάρχουν σε εσά να βοηθήσουν και εμάς και τα Νάπαλιν. Και επανέρχομαι σε αυτήν την εικόνα που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλής. Υπάρχει ανάγκη να δημιουργήσουμε μια γέφυρα ανάμεσα στην υπηρετική Ευρώπη και στα κράτη του Καριφόρουμ, να κάνουμε μια γέφυρα πάνω από τον Ατλαντικό. Θέλουμε λοιπόν μια γέφυρα που δεν θα επιτρέπει μόνο την κυκλοφορία, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Χρειάζεται και δράση, ταλέντο, πολιτική βούληση και πάνω απ' όλα ενεργοποίηση. Ο Μάρκ Ταραμπέλα. Έχω και μια απορία γιατί χθε είδα ένα ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω αν ήταν αξιόπιστο. Ε, άκουσα ότι η, ο αμπελοϊνικό τομέας θα εκλείψει λόγω της αύξησης θερμοκρασίας, Γιατί αν αυξηθεί η θερμοκρασία κατά 2-2,5 βαθμούς ή ίσω το Βέλγιο γίνει μεγάλη α, είναι ο παραγωγό χώρα. Γιατί το 1700 και ε, οι κάτοικοι τη Βουργουνδία ξερίζωσαν τα μπέλια μας στη λίγη. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν λόγω της αύξησης θερμοκρασία να επηρεαστεί η τοπική γεωργική παραγωγή που είναι κέρια για τον οικονομικό σα κλάδο. Υπάρχουν μελέτες που έχουν γίνει ενδεχομένω από τους γεωπόνους σα για το πώς θα επηρεάσει το μέλλον αυτή η υπερθέρμανση του πλανήτη τη γεωργική παραγωγή. Σα ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, βεβαίω και θα την επηρεάσει στην Καραϊβική Έχουμε ελάχιστα συστήματα άρδευσης των καλλιεργειών. Και οι προβλέψεις λένε ότι οι... Ε, πολλές φορές θα έχουμε τις βροχοπτώσεις που θα έχουμε σε 20 λεπτά τις βροχές ολόκληρου του έτους. Και δεν θα υπάρχει δυνατότητα ε, λόγω του κόστους της άρδευσης και της έλλειψης πρόσβασης σε συστήματα ε, γλυκού νερού να συνεχίσουμε να έχουμε την παραδοσιακή μας γεωργία, μια και δεν θα μπορούμε καθόλου να αρδεύουμε τις καλλιέργειες. Και υπάρχει και ένα άλλο ζωτικό θέμα του τουρισμού, γιατί ο τουρισμός είναι ε, βασικός πλουτοπαραγός κλάδος σε πολλά νησιά. Και ο τουρισμός τροφοδοτεί τις οικονομίες σχεδόν των περισσότερων χωρών της Καραϊβικής. Οπότε δεν είναι μόνο η γεωργία που θα επηρεαστεί, αλλά και ο τουρισμός. Είπατε να δημιουργήσουμε γέφυρες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καραϊβικής. Μα ήδη έχουμε η Μαρτινίκα, 70 ε, μίλια από την Αγία Λουκία και η Γουαδελούπη ελάχιστα μίλια από την Αντίγουα. Οπότε ε, είμαστε και συνδεδεμένα μέλη της Κάρικομ, χώρες της Ανατολικής Καραϊβικής και υπάρχει δυνατότητα της εμβάθυνσης των περιφερειακών δεσμών, όχι μόνο των πολιτιστικών, γιατί έχουμε ε, ίσως κάποιες ιστορικούς διχασμούς, αλλά είμαστε ενωμένοι και ίσως ε, χρειαζόμαστε περισσότερες ε, ενέργειες, γιατί κάποιες, ε, κάποιοι φόροι στο Ρούμι, για παράδειγμα, στην Καραϊβική δημιούργησαν φραγμούς και στα αγαθά και στις υπηρεσίες πολλές φορές. Και γι' αυτό θα ήθελα, μια και επίκυνται οι διαπραγματεύσεις για το περιφερειακό πρωτόκολλο, να συζητήσουμε τη μείωση ενδεχομένω αυτών των φραγμών, ώστε να αξιοποιήσουμε καλύτερα την παρουσία της Ευρώπης και στην Καραϊβική. Σας ευχαριστούμε που μας υπενθυμίσατε, Δ. Ισμαήλ, ότι τα υπερπόντια διαμερίσματα, τα γαλλικά υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα είναι η πρώτη πύλη της Ευρώπης ε, με γεωγραφική και ιστορική εγκύτητα με τις χώρες του Καριφόρου. Και έχουμε και εδώ πολλά θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτηση και επεξεργασίας. Και περάσατε και στο επόμενο θέμα της ε, συνεδρίασης, της ανάγκης ε, σφαιρικής προσέγγισης και στις διαπραγματεύσεις για την περίοδο μετά το Κοτονού. Αυτό θα συζητήσουμε τώρα και εξοχότατη ε, Σέιλα Σιλιμόντε, κυρία πρέσβυρα. Είστε πρέσβυρα της ε, Τζαμάικα, αλλά και συντονίστρια των κρατών της Ανατολικής Καραϊβικής ε, στις Βρυξέλλες. Οπότε εκπροσωπείτε το σύνολο των κρατών της Καραϊβικής κατά κάποιο τρόπο. Και είναι σημαντικό να σας ακούσουμε σήμερα για το τι γνώμη έχετε για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις και τι ανάγκες έχετε τι επίγουσες ανάγκε έχετε ε, στις διαπραγματεύσει αυτές και που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και από εμά. Καλώς ήρθατε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Έχω την τιμή να απευθύνομαι στο Σεβαστό Ακροατήριο εκ μέρους των 12 πρεσβειών που εκπροσωπούν τα 16 κράτη ε, της ομάδας των χώρων Καραϊβικής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που ε, επιδεικνύεται στις υποθέσεις Καραϊβικής και στις, ε, α, στην ανάγκη να υπάρξουν σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο περιοχών. Έχουμε ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία μετά το Κοτονού μια ευκαιρία να ενδυναμώσουμε τη σχέση μεταξύ της Ένωσης και των χωρών ΑΚΕ. Θέλουμε να εμβαθύνουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών ΑΚΕ και να συγχρονίσουμε τη βάση για την ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων στο πλαίσιο του θεματολογίου 2030. Από τότε που στορμολογήθηκαν οι διαπραγματεύσει, εκπρόσωποι τη Καραϊβική ε, συμμετείχαν εξ ολοκλήρου σε όλε τι πτυχέ τη προετοιμασία και τη εξαγωγή τη όλη αυτή διαδικασία για να τεθούν τα θεμέλια τη συζήτηση ε, του πρωτοκόλλου και συμφωνία σε υπουργικό επίπεδο. Και λαμβάνουμε υπόψη ε, και τη συνεισφορά όλων των φορέων τη περιοχή. Νομίζω ότι στις ε, διαπραγματεύσεις ε, ε, συμφωνούμε όλοι ότι έχουν επιτευχθεί σημαντικές πρόοδοι μέχρι τώρα. Έχουμε σταθεροποιήσει το κείμενο και τους τίτλους σημαντικών μέρων αυτής της συμφωνίας. Βέβαια υπάρχουν ακόμη κάποιες διαφωνίες και θα γνωρίζετε ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση των επικεφαλής διαπραγματευτών υπήρξαν κάποιες ρυθμίσεις και διακανονισμοί για να λυθούν αυτά τα ζητήματα τις επόμενες εβδομάδες. Η Καραβική θα συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο της σε συνεργασία συνεργασία με του εταίρου μα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών ΑΚΕ, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει, ελπίζουμε, μέω στα τέλη του Απριλίου. Καρεβική, κύριε Πρόεδρε, είναι δεσμευμένη στην αρχή τη σύναψη μια ενιαία συμφωνία που θα εδράζεται στο κεκτημένο του Κοτονού. Ε, συμφωνούμε με το στόχο να έχουμε όριμε σχέσει, να είμαστε εταίροι ισότιμοι και να εργαζόμαστε μαζί για να προωθήσουμε το πολυμερέ σύστημα στην επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων. Βιώσιμη ανάπτυξη, βέβαια, είναι η βασική μα προτεραιότητα. Βεβαίω, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στην περιοχή μα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των διατάξεων τη συμφωνία και ιδίω στο περιφερειακό πρωτόκολλο. Έχουμε γνωστά τροτά σημεία τα οποία επηρεάζουν το ρυθμό και τη βιωσιμότητα της ανάπτυξής μας. Ε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ε, βλέπουμε ότι υπάρχει η ενδεικτική δομή ε, περιφερικής εταιρική σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών. Οι διαπραγματεύσεις συζήτησαν τα θέματα της κοινωνικής συνοχής, ανθρώπινων δικαιωμάτων, ειρήνης, ασφάλειας, διακυβέρνησης, τρόπινης ανάπτυξη. Έχουμε λοιπόν σταθεροποιήσει κάποιο σώμα κειμένου και έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσει για την αλληλέγγυα ανάπτυξη ανάπτυξη και μεγέθυνση και ε, θα δούμε και τα άλλα τα ζητήματα άμεσα. Υπάρχουν και κάποια ζητήματα, ε, δεν μας ε, εκπλήσει αυτό. Περιλαμβάνουν για παράδειγμα τις ανησυχίες μας για την αντιμετώπιση της φορολογίας και των διεθνών επιχειρηματικών υπηρεσιών αν υπάρχει αυτή η νέα συμφωνία ε, οικονομικής εταιρικής σχέση, ανησυχούσαμε πω υπάρξουν προβλήματα ε, στι συναλλαγές μα και θέλουμε νέα συμφωνία να διευκολύνει τι χώρε μα να μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τι εμπορικέ και άλλες διατάξεις της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης. Ε, θέλουμε επίση να υπάρχει μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην ανάπτυξη, στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα είναι στον το πιο προοδευτική και στα ζητήματα που άπτονται τη μετανάστευση. Ελπίζουμε να βελτιώθει η δημιουργία υποδομών, μεταφορά τεχνολογία για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και ιδίω ε, τη νέα γενιά. Θέλουμε επίση να υπάρξει μεγαλύτερη περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και οι βασικοί οικονομικοί φορεί να μετασχηματιστούν, ε, να δημιουργηθεί, ε, να δοθεί έμφαση στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών και κλάδων, στον τομέα του πολιτισμού θα δούμε ποιε θα είναι οι τελικέ διατάξει τη συμφωνία. Ελπίζουμε ε, να αντικατοπτρίζει τη σημασία ε, που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι χώρε σε αυτήν την εταιρική σχέση. Οι βασικέ μα ανησυχίε ε, παραμένουν στο ότι θα πρέπει όταν καταρτήσουμε μια νέα εταιρική σχέση να έχουμε τη δυνατότητα ω χώρε ΑΚΕ να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών μα. Και Υπάρχει και υπάρχουν και οι στόχοι, μια σύνοψη των στόχων και για τα περιφερειακά πρωτόκολλα. Πρώτον, ε, θα πρέπει να έχουμε την βασική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Καραϊβικής που θα προωθήσει βασικούς στόχους Επίσης έχουμε την EPA, ε, ε αυτή την οικονομική εταιρική σχέση που δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο άλλες δεσμεύσεις. Επίσης θέλουμε περιφερειακή συνεργασία και ένταξη, αλλά να αναγνωριστεί ταυτόχρονα ε, ότι υπάρχουν και διαφοροποίησεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και τέλος θα πρέπει αυτή η νέα συμφωνία να ενισχύει στην οικονομική, περιβαλλοντική κοινωνική αφεκτικότητα των ευάλωτων οικονομιών της Καρεβικής. Επίσης θα πρέπει να δοθεί στήριξη στην IT ε, που είναι μία από τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και θα πρέπει να υπάρχουν ε, συγκεκριμένες διατάξεις στα περιφερειακά πρωτόκολλα που θα καλύπτουν ε, τις ανάγκες αυτής της χώρας και εκτόν έχουμε την ανάγκη να έχουμε μια νέα συμφωνία που θα λαμβάνει υπόψη και τις φιλοδοξίες των χωρών της Καραϊβικής προς ανάπτυξη. Είναι μια προσπάθεια μακρόπνοη και πολύ ελπιδοφόρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, εξοχότατη. Πραγματικά ήταν πολύ βαρισίμαντη η ομιλία σας και νομίζω ότι η ανάπτυξη μόνο χωρίς αποκλεισμούς νοείται και δεν θα κουραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε και με τη βούληση να αλλάξουμε την καθημερινότητα, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, θα πρέπει να συνεργαστούμε οπωσδήποτε και να μην αποκλείουμε κανέναν. Μιλήσατε για κινητικότητα, για ανθεκτικότητα, εξαιρετικά σημαντικά θέματα όλα αυτά. Θα ήθελα τώρα να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την εποχή μετά το Κοτονού. Φρανσουά Ρουντιέ, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Χαιρόμαστε και πάλι για την ευκαιρία που έχουμε για ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους πρέσβεις ε, και τα μέλη της αντιπροσωπείας. Εγώ δεν χρειάζομαι τρία λεπτά. Προτιμώ να αφήσω λίγο χρόνο στο συνάδελφο Ντενή, που έχει και αυτός κάτι να σας πει. Χαιρόμαστε αρκετά από την πορεία των διαπραγματεύσεων και συμμερίζομαι ε, την ανάλυση που έκανε για την κατάσταση η πρέσβης Μόντε. Γενικώ έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε τα μισά κεφάλαια. Τα υπόλοιπα μισά είναι εκρεμή, αλλά μερικά στοιχεία είναι ήδη γνωστά. Κάποια σημεία δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά αφορούν το κοινό σημείο. Αλλά γνωρίζουμε την άγουσα που θα ακολουθήσουμε και έχουμε επίγνωση ότι έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας, με μια πολύ φορτωμένη δουλειά σε αυτό το χρόνο, αλλά πιστεύω ότι θα πατήσουμε τον γκάζι και θα ε, ολοκληρώσουμε έγκαιρα τη συμφωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του πρωτοκόλου για την Καραϊβική. Θα πρέπει φυσικά να δούμε τα ευάλωτα σημεία της περιοχής ε, και αφιερώσαμε 35 λεπτά στη συζήτηση της βασικής ευπάθειας που επηρεάζει όμως και τις υπόλοιπες γιατί οι κλιματικές αλλαγές ενισχύουν όλα τα υπόλοιπα ευάλωτα σημεία των χωρών ε, της Καραϊβικής λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα, του μικρού μεγέθους της οικονομίας, ε, των ε, κοινωνικών ευπαθειών, θέματα επιμελητίας, περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής και ούτω καθεξής. Για μας το πλαίσιο μετά την Συμφωνία Κοτονού και το πλαίσιο για το πρωτόκολλο της Καραϊβικής θα μας χρησιμεύσουν για να δημιουργήσουμε μια πραγματική συμμαχία, μια ουσιαστική εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, χωρών αυτών για να, για να ξεφύγουμε από αυτή την παλιά σχέση δωρητή και δικαιούχου που είχαμε στο παρελθόν. Γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε από κοινού σε συνεργασία, στα πλαίσια μια συμμαχία και κυρίω στα θέματα πολυμέρειας, γιατί η πολυμέρεια απειλείται παγκοσμίω. Και η κλιματική αλλαγή είναι ένα παράδειγμα, γιατί είχαμε ένα ολόκληρο σύστημα για τις ε, πολιτικές μας, οπότε θα πρέπει να συνεργαστούμε για να προστατεύσουμε την πολυμέρεια και στα θέματα του διεθνούς εμπορίου. Αναφερθήκατε στην διακυβέρνηση των ωκεανών επίσης και για αυτά τα θέματα θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και για τις πολιτικές κρίσεις επίσης. Όπως είπατε λοιπόν, ε, θα πρέπει με μεγάλη φιλοδοξία, πολλή θέληση και αποφασιστικότητα με πυγμή να προχωρήσουμε και ταχαίως και νομίζω ότι συνεργαζόμαστε πολύ καλά με τους συναδέλφους μας. Χαίρομαι με τόση σύγκληση και σύμπνοια δημιουργείται μεγάλη αισιοδοξία ε, ότι θα τελεσφορήσουν οι διαδικασίες και μάλιστα εμπρόθεσμα παρόλο που το χρονοδιάγραμμα μας πιέζει κάπως. Και η συνάδελφος σημειώνει πυρετοδός όλα αυτά τα σημεία, γιατί υπάρχουν πραγματικά πολύ θεμελιώδη ζητήματα. Ο παρακαθήμενός σας είναι ο Ντενίτσα Λάν από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Θα ήθελα να μας πει και εκείνος δυο λόγια για να εκμεταλλευτούμε και τη δική του εμπειρογνωσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι καλύφθηκα σχεδόν όλα τα σημεία. Επιτρέψτε μου να επιμείνω και από πλευρά μα σε αυτό που είπε ο συνάδελφος, στο γεγονός ότι το έργο που κάνουμε στα πλαίσια της εποχής μετά το Κοτονού και τη συμφωνίας μετά το Κοτονού θα μας επιτρέψει να σφυριλατήσουμε ακριβώς αυτό το σύγχρονο συνασπισμό, αυτή τη σύγχρονη συμμαχία μια σύγχρονη εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών τη Καραϊβική. Και αυτό το περιφερειακό πρωτόκολλο για την Καραϊβική θα είναι πολύ σημαντικό και θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε αυτή τη βάση για τη συμμαχία μας. Επανειλημμένως αναφερθήκατε στο θέμα της σύγκλησης των απόψεων. Είναι σαφές ότι για όλα αυτά τα θέματα υπάρχει πραγματική σύγκληση. Υπάρχουν πολλές κοινέ ιδέες και προτάσεις και χαιρόμαστε ιδιαίτερος που συμμετέχουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αναφερθήκαμε στις κλιματικές δράσεις, στα διάφορα ευάλωτα σημεία, στις ευπάθειες που έχουν οι χώρες αυτές, στο θέμα της περιφερειακής ολοκλήρωσης που είναι επίσης σημαντική και οικονομική ολοκλήρωση με τις μελλοντικές συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Και όπως αναφερθήκατε και εσείς, Πρόεδρε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την, και την κυκλική οικονομία ή την πράσινη οικονομία ή τη γαλάζια οικονομία, όπως την αναφέρουμε, για τους ωκεανούς. Επίσης, ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό στη συζητήση με τους εταίρους μας από την Καραϊβική είναι το θέμα και το έργο μας για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα μας επιτρέψουν να βάλουμε τα θεμέλια των μελλοντικών μας δράσεων και κυρίως ε, να δούμε και τι μορφή θα έχει ο τελικός μηχανισμός. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ε, για τα θέματα αυτά, γι' αυτό δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα. Πάντως, για τις προθεσμίες ελπίζουμε ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αν μη τι άλλο ένα προσχέδιο συμφωνίας που θα ακολουθήσει την πορεία του γιατί ο δρόμος ε, στη συνέχεια θα είναι και πάλι μακρύς. Σας ευχαριστώ πολύ. Είδα να μη διούν οι εταίροι, οι προσκεκλημένοι μας σε ό,τι αφορά τη φιλοδοξία και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Ε, σας ευχαριστώ για τι πληροφορίες και σας ευχαριστώ και για την ιδέα αυτή τη σύγχρονη εταιρική σχέση που αναφέρατε, γιατί ίσως ε, και εδώ θα πρέπει να δούμε ε, πώς αυτή η φιλοδοξία μας μπορεί να μεταφραστεί σε πράξη, να συγγράψουμε διαφορετικά αυτή τη συμφωνία, να μην έχουμε ένα copy-paste κάθε φορά, αλλά να δούμε ε, και να διερωτηθούμε. Κάνουμε τα πράγματα ως συνήθως και τελικά πάντα με το ρίσκο της αποτυχίας, διότι έχουμε νέα προκλήσεις, νέες κατεπίγουσες περιστάσεις. Ε, δεν θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Ε, νομίζω ότι έχουμε την ευθύνη να συνοικοδομήσουμε το μέλλον μας. Νομίζω τώρα ότι Καλό θα ήταν να, ζητήσω από τους συναδέλφους που θα ήθελαν το λόγο και μετά να κλείσουμε η Μαρή Πιέρ Βεντρέν. Ίσως για να μας πει δύο λόγια γνωρίζω πόσο ε, σας ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα. Είστε προσιλωμένοι και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Στεφάν. Ε, καλησπέρα σε όλες και όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την μαρτυρία σας πρώτα απ' όλα που πραγματικά ενσαρκώνει την πραγματικότητα και ήταν πολύ σημαντικό να ακούσουμε διαστόματό σας ε, την μαρτυρία Μενιουέλ Μακρόν και η Γαλλία όπως ξέρετε αγωνίζεται η Συμφωνία των Παρισίων αποτελεί σημείο αναφοράς και σημαντική ρήτρα στι ε, συμφωνίε. και το βλέπουμε για τις διαπραγματεύσεις για το μετά το Κοτονού ότι επιμένουμε να είναι στο επίκεντρο η Πράσινη Συμφωνία ε, η Γκρέτα Τούρμπερκ στο Κοινοβούλιο και γενικώ υπάρχει αυτή η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Και η συμφωνία θέλουμε να είναι μια ρήτρα σημαντική ε, στο πλαίσιο της συμφωνίας. Θεωρείτε ότι είναι πιθανό αυτό και τι έχετε να πείτε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Να σας πω ότι μας, ε, μας μένει ένα πεντάλεπτο πριν το τέλος ε, θα τα λύσει απόψε. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να είστε πολύ σύντομοι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που εκφράσετε την εκτίμησή σας στο έργο που κάνουμε και στη σημασία που αποδίδει τη κλιματική αλλαγή. Ε, το θέμα του κλίματος που επηρεάζει όλες τα συμβαλόμενες πλευρές σίγουρα αναγνωρίζεται και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη δική μας πλευρά. για να γνωρίζετε από τις διάφορες χώρες και τις ε, διάφορες ε, ε, ομάδες χωρών, νησιωτικές, περίκλειστες κτλ. Διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές εμπειρίες σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Αλλά όλοι συμφωνούμε, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα η κλιματική αλλαγή. Και φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει και τα ζητήματα από τότε της διακυβέρνησης των ωκεανών με την ανάγκη να ληφθούν μέτρα μετριασμού και κάτι άλλο που δεν αναφέρθηκε και είναι πολύ σημαντικό παρόλα αυτά είναι η κλιματική χρηματοδότηση που είναι κομβικό σημείο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων μας και πρέπει να δούμε ποιο είναι το πακέτο, ποια είναι η δέσμετρο που θα εγκριθεί εν τέλει. Ελπίζουμε όμως να μπορέσουμε ήδη ε, να εκταμιεύσουμε τα κονδύλια που ήδη είναι πολλά και για το περιφερειακό πρωτόκολλο σίγουρα υπάρχουν δράσεις που μπορούν να ληφθούν ε, για την ανάπτυξη των οικονομικών κλάδων και στον τομέα του πολιτισμού ακόμα και της ε, περιβαλλοντικής προστασίας των τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς, των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλα αυτά τα ζητήματα επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Άρα δεν υπάρχει καμία αφιβολία πως είναι στο επίκεντρο, είναι στην πρώτη γραμμή και θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους του θεματολογίου του 2030. Και το κλίμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο ε, με όλους αυτούς, τουλάχιστον όχι όλους τους περισσότερους από αυτούς τους στόχους. Σίγουρα θέλουμε να επιδείξουμε τη δέωσα φιλοδοξία και σίγουρα η Συμφωνία των Παρισίων είναι σημείο αναφοράς. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω με την αποφασιστικότητα και την καρηγορηματική σας ε, αυτή απάντηση θέλουμε να σας χειροκροτήσουμε. Έτσι αυτό βγαίνει αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ ε, που δίνετε σε όλα αυτά τα θέματα σημασία. Εξοχότητε, ε, δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς να δώσετε κάποια σχόλια. Όχι. Αντί να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες από τις κάλυψε τέλεια η πρέσβυρα, θα ήθελα να πω ότι από τις 16 κράτη-μέλη του Καριφόρουμ έχουμε εκπροσώπους από 15 χώρες εδώ σήμερα και άλλους τέσσερις ε, ε, πρέσβεις πέραν του υποφαινομένου και της πρέσβυρας της Τζαμάικα. Κάτι που δείχνει πόσο σημαντικές είναι οι ανταλλαγές απόψεων. Και σας ευχαριστώ για τον ηγετικό σας ρόλο, σας ευχαριστώ για το ρόλο της αντιπροσωπής σας, γιατί πραγματικά αναζωογονείτε έχετε αναζωογονήσει του τελευταίου μήνε το έργο αυτή τη αντιπροσωπεία και προσβλέπουμε στην ε, συνάντηση του Μαρτίου. Και ό,τι μπορούμε εμεί ω πρέσβει ε, του Καριφόρουμ να κάνουμε, πείτε μα και θα το κάνουμε. Σα ευχαριστώ θερμότατα, πραγματικά, ειλικρινά σα λέω. Σα ευχαριστώ για την εμπειρογνωμοσύνη σα και ε, μερικέ φορέ είναι δύσκολο μόνοι μα να έχουμε κατάλληλη άποψη της κατάστασης της χώρας Καλιφόρουμ. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε και την δική σας άποψη, γιατί εσείς ε, είστε εξοικειωμένοι με την κατάσταση επιτόπου και μας χρειάζεται και η δική σας κοπιά. Έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτή τη συμφωνία και να την εμπλουτίσουμε με συγκεκριμένες δράσεις, γιατί είναι σημαντική και για τις δύο πλευρές. Θέλουμε μια αμοιβαίως υποφελή συμφωνία στα πλαίσια μιας σύγχρονης εταιρική σχέσης, όπως πολύ εύγλωτα μας είπαν ε, εδώ οι καλεσμένοι μας. Και θα πρέπει να καινοτομήσουμε και να προσφέρουμε λύσεις και στα πλαίσια της γαλάζιας οικονομίας. Στις 23 Μαρτίου θα έχουμε μια πολύ σημαντική στιγμή για την αντιπροσωπεία του Καριφόρουμ, γιατί θα έχουμε τη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή και θα είναι όλοι παρόντες εκεί. Η ευρύτερη οικογένεια του Καριφόρουμ ε, θα βρίσκεται σε πλήρη σύνθεση στη συνεδρίαση εκείνη τη 23 η Μαρτίου, γι' αυτό και θα πρέπει να προετοιμαστούμε και μάλιστα σε λίγο θα έχω τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό μου από το Καριφόρουμ για να προετοιμάσουμε από κοινού την επόμενη συνεδρίαση της 23, ης Μαρτίου και στις 15 Ιουνίου, 3 ε, η ώρα στις Βρυξέλλες, θα ξαναβρεθούμε στα πλαίσια της δικής μας αντιπροσωπείας του Καριφόρουμ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ραντεβού τη Δευτέρα με κάποιους από εμά και σας ευχαριστώ γιατί περάσαμε πραγματικά πολύ πλούσια και καλή στιγμή. Καλή σας βδομάδα και ευχαριστώ και τους διερμηνείς Λεοπρόεδρος και τη Γραμματεία.